Τροπολογία 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 Μανομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 αντί με κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 58 μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 61, μονομαστική κλίση, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Άρθρο 1685 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά στο επαληθεύσουμε και ηλεκτρονικά. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Παράγραφος 35, τέτερα, τέ, τέσσερα τμήματα, μονομαστική κλίση, πρώτο τμήμα, άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πρώτο τμήμα 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 5 με πρώτο τμήμα άρτη ψηφοφορία, παράγραφος 52. Πέρας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα άρτη Πέρας. Εγκρίνεται. 24 μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 60, αρχικό κείμενο, μονομαστική κλίση, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 63, αρχικό κείμενο, μονομαστική κλίση, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 64 σε τρία τμήματα, το αρχικό κείμενο πάντα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παραγράφος 65 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 67 αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 68 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 πέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο Μονομαστική κλίση άρθρη ψηφοφορία. Ακαταπίπτει, συγγνώμη, ο πρόεδρος. Τροπολογία 26 τώρα μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο. Μονομαστική κλίση. Α, καταπίπτει. Καταπίπτει, λέει ο πρόεδρος. Καταπίπτει και αυτό. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο. Μονομαστική κλίση. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Το κείμενο εγκρίνεται. Παράγραφος 75, τροπολογία 27, μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφο 77 αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 28, μονομαστική κλίση, άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Το κείμενο απορρίπτεται. Τροπολογία 29, πρώτο τμήμα υπέρ κατά Υπέρ παρακαλώ, σηκώστε το χέρι σα Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με κλίση, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο με κλίση, άρτη ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Κατά το αρχικό κείμενο, πάμε στην παράγραφο 83 υπέρ κατά. Σηκώντε το χέρι υπέρ της 83 κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Το κείμενο εγκρίνεται. Παραγράφος 106, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Την 90 τη ξεχάσαμε. Ονομαστική κλίση ψηφίζουμε τροπολογία 90. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 106, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 πονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 91 και έχουμε πολλές τροπολογίες ακόμα. Να σηκώνετε το χέρι σας παρακαλώ πολύ, γιατί βολικά θα κάνουμε συνεχώς επαληθεύσεις. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 2. Πολύ ωραία. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68 Πολύ ωραία. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 67. Άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Έχουμε 100 ακόμα τροπολογίε. Σα το υπενθυμίζω απλώ. Πέρα. Εγκρίνεται. «68 υπέρ» «κατά» «αποχές» «απορρίπτεται» Πολύ ωραία. Ηλεκτρονική επαλήθευση, τροπολογία 68. Αλλά να σηκώνετε το χέρι σας, γιατί μου είναι αδύνατο να καταλάβω την πρόθεση ψήφου. Πέρας. Απορρίπτεται. 30 με ονομαστική κλίση άρτε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 31. Μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32. Μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρασε Εγκρίνεται. Παράγραφος 173, δύο τμήματα, μονομαστική κλίση και τα δύο άρτη ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Πέρασε. Εγκρίνεται το κείμενο. Δεύτερο τμήμα, μονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 33 τώρα, μονομαστική κλίση, ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 209 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 214, με ονομαστική κλίση ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος, μάλλον τροπολογία 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 219 υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο επαληθεύσουμε και ηλεκτρονικά. Ψηφίσουμε παρακαλώ. Πέρασε. Απορρίπτεται. Παράγραφος 223, τροπολογία 10, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται 97, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται 93, υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο επαληθεύσουμε και ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Ναι, ναι, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ναι, ναι, κοντρόλο ε, λέμε στα Ιταλικά. Το ελέγχουμε δηλαδή ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Να. 35 με ονομαστική κλίση. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 250. Υπέρ. Κατά. Δεν ψηφίσει κανείς όμως πια, έτσι δεν είναι. Υπέρ της παραγράφου 250, παρακαλώ, αρχικό κείμενο. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 μονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 263, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, αγκρίνεται, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά σε παληθεύσουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 263. Πέρασε. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 δίμα ονομαστική κλίση ψηφίζουμε Πέρας. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 76. Μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ελεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 77. Ψηφίζουμε. Πέρασε εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 79 με ονομαστική κλίση ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 94 ονομαστική κλίση. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 304, τροπολογία 21, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική επαλήθευση για 95 πολύ ωραία ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται είχατε δίκιο 96 σε δύο τμήματα και τα δύο μονομαστική κλίση ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα Πέρασε. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Το κείμενο εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι επόμενες και φτάνουμε στη 42 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά Υπέρ τη 16 παρακαλώ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε για τροπολογία 81 με ονομαστική κλίση. Απορρίπτεται. Παράγραφος 326, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 333. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 345 μονομαστική κλίση άρθρη ψηφοφορία. Να ελέγξουμε τι ακριβώς τώρα. Τροπολογία 82. Πολύ ωραία. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά τροπολογία 82. Άρχιτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Μονομαστική κλίση τώρα ψηφίζουμε την παράγραφο 345. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 347. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 μονομαστική κλίση ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 359 μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 368, ψηφίζουμε ονομαστική κλίση. Πέρασε. Το κείμενο εγκρίνεται. 45 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 45, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48. Μονομαστική κλίση ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 53D, μονομαστική κλίση ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 401, άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 54 D ονομαστική κλίση ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία ντύμα, ονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Καλησπέρα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 49 υπέρ. Κατά. απόχέ. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Με ονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18, ονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Παράγραφος 408. Το αρχικό κείμενο μονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 409. Άρτη ψηφοφορία, μονομαστική κλίση. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50 με ονομαστική κλίση άρθρη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος, μονομαστική κλίση, άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Το κείμενο εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Κόφοτ και Νέντερμαϊερ. Σίγουρα άξιζε το χειροκρότημα όχι μόνο για το περιεχόμενο τώρα τη έκθεση αυτή, αλλά και για το ότι είχαμε μια πολύ μακρά ψηφοφορία. Περνάμε τώρα στην έκθεση Φροντζούλικα Θεσμική Συμφωνία Πλαίσιο Ευρωπαϊκή Ένωση Ελβετία, τροπολογία 1, μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3, μονομαστική κλίση, ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρο... Πολύ ωραία. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της α, τροπολογίας αυτής, άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά ποχέ. Εγκρίνεται. Η σύσταση στο σύνολό της μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Το κείμενο εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Φουντζούλικα. σας ψήφου τώρα. Παρακαλώ όσοι εγκαταλείπουν την αίθουσα να το κάνουν αθόρυβα για να μπορέσουμε να περάσουμε στις αιτιολογικές, ε, στις αιτιολογίες ψήφου απρόσκοπτα. Περνάμε λοιπόν στις αιτιολογήσεις ψήφου. Ξεκινάμε με την έκθεση κυρίας Ούλσκοκ για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας. Η κυρία Άλεξ Μάγερ είναι η πρώτη. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα την έκθεση. Δεν έχω πρόβλημα με τις εποχικές αλλαγές της ώρας και πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε διπλή θερινή, δηλαδή να έχουμε μία επιπλέον ώρα το καλοκαίρι. Γιατί αν μεταφέρουμε τις ώρες με ήλιο, προ, φως προς το τέλος της μέρας, θα εξοικονομήσουμε και ηλεκτρική ενέργεια και εκπομπές άνθρακα και θα διευκολύνουμε και τις τουριστικές δραστηριότητες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ρολόγια που χτυπάνε, 5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν υπογράψει την αίτηση κατά του Brexit. Να σταματήσουμε το ρολόι. Έχουν σπάσει στο σελίδες ε, της Βρετανικής Βουλής. Να σταματήσουμε λοιπόν το ρολόι του άρθρου 50. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δρογεύσκη. Εδώ και μερικά χρόνια είμαι διακαής ε, υπέρμαχο ε, τη μη εποχική αλλαγή ώρα, ούτε προ τη χειμερινή, ούτε προ τη θερινή ώρα. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν πολλές διαταραχές από αυτή τη διπλή αλλαγή ε, ώρας από τη χειμερινή προς τη θερινή και αντίστροφα. Χρειάζεται λοιπόν κάποια εναρμόνιση. Αυτό είναι προφανές. Και επίσης μια μεταβατική περίοδος για να προσαρμοστούμε στην κατάσταση. Η τα παρούσα όμως πρόταση το, της προθεσμίας της 18 μήνης παρά είναι μακρά μεταβατική περίοδος. Τι νόημα έχει ε, κάτι τέτοιο. Δείχνει έλλειψη ετοιμότητας ε, για άμεση δράση εκεί που χρειάζεται πραγματικά και αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει ε, σχετικά γρήγορα. Θα ήθελα λοιπόν να σταματήσει η εποχική αλλαγή της ώρας και το πολύ να προβλέψουμε μεταβατική περίοδο 12 μήνη και όχι 18 μήνη όπως προτείνεται κυρία Βάουτμας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης, υπέρ της κατάργησης ε, της ετήσιας αλλαγής ε, ώρας ε, και ψήφισα υπέρ της διατήρησης της θερινής ώρας. Γιατί, Γιατί και οι πολίτες μας θέλουν βεβαίως να υπάρχει μία ώρα και θέλουν να υπάρχει η θερινή ώρα και πρέπει να γίνεται στο δυνατό. Ήλπιζα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα είχαμε την τελευταία αλλαγή της ώρας, αλλά η έκθεση ε, και το Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι χρειαζόμαστε χρόνο. Χρόνο να υπάρξει ένας μηχανισμός ε, συντονισμού ότι ε, βεβαίως όλα αυτά ε, είναι ζητήματα που αφορούν και την οικονομία και την ιστορική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είμαι ικανοποιημένη με αυτήν την ώρα και ελπίζω 2021 ε, να αλλάξουμε ώρα μια και καλή και να πάμε στη θερινή ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω την κυρία Αγγιλέρα στην αίθουσα. Αποσιάζει. Οπότε περνάμε στην κυρία Σούιτσα για να αιτιολογήσει την ψήφα της. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι η εποχική αλλαγή της ώρας δύο φορές το χρόνο επηρεάζει αρνητικά και την υγεία και την κυκλοφορία, το ενεργειακό σύστημα, τη γεωργία. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν τάχθηκε πέρ της κατάργησης εποχικής αλλαγής της ώρας. Αν και θα προτιμούσα να μην περιμένουμε ε, το 2020 ε, να, να μείνουμε από τώρα στη θερινή ώρα. Είμαι κατά τέτοιες ε, ε μεταβατικές περίοδου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μείνουμε στη θερινή ώρα. Και οι μελέτες άλλωστε έχουν δείξει και αποδείξει ότι η μεγαλύτερη υποστήριξη φέρει η θερινή ώρα. Θα υπάρξει πρόβλημα όμως στο συντονισμό, από ό,τι φαίνεται. Θα πρέπει λοιπόν να συνεννοηθούμε ε, γιατί αν ε, εφαρμοστούν διαφορετικές ώρες στα διάφορα κρατημέλη, τότε είναι που θα έχουμε αρνητικές επιπτώσεις στις, ε, στις διασυνοριακές μετακινήσεις. Νομίζω ότι η πιο δόκιμη αλλαγή είναι υπέρ της θερινής ώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σέινφελτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το θέμα και πολλές πρακτικές συνέπειες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, ε, γιατί δύο φορές το χρόνο αλλάζουμε το ρυθμό της ζωής μας, αλλάζοντας ε, την ώρα στα ημερολόγια μας και στα ρολόγια μας. Αυτό επηρεάζει ε, τις μεταφορές, τον τουρισμό, την οικονομία, τους επιχειρηματίες και γι' αυτό είμαι υπέρ της κατάργησης της εποχικής αλλαγής. Αλλά έχω πολλές αμφιβολίες και ενδιασμούς. Γι' αυτό και κάνω έκκληση για να δούμε πώς θα υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Νομίζω ότι είναι μια ριζική κατάργηση άμεση πολύ προβληματική. Επίσης υπάρχει πιθανότητα ακόμη και μετά την κατάργηση των εποχικών αλλαγών να έχουμε διαφορετικές ώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή κάθε κράτος θα επιλέξει διαφορετική ώρα για να εφαρμόσει. Αυτό είναι ακόμη πιο επικίνδυνο. Κύριος Χάναν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η συνάδελφο εδώ πέρα μιλάμε για την αλλαγή τη ώρα και μα είπε να σταματήσουν τα ρολόγια του Brexit. Δηλαδή, αν ε, γίνουν τελικά ευρωεκλογέ, ε, δεν φαντάζομαι να έρθουν πολλοί ε, εργατικοί ευρωβουλευτέ. Κι όμως όλοι πλέον το θεωρούν δεδομένοι ότι είναι πλέον ευρωπαϊκή αποφασία. Ακόμα και το σε ποια χρονική ζώνη βρίσκεται κάποιο. Δεν είναι υπόθεση των κρατών μελών. Δηλαδή εγώ θεωρώ, μπα, αν θέλετε την άποψή μου, ότι θα έπρεπε να έχουμε μονίμως την ε, θερινή ώρα, γιατί αντικατοπτρίζει ακριβώς το σύστημα αυτό τον τρόπο εργασία τη προηγούμενη γενιά. Αλλά είναι ένα περίεργο σχολείο για το πώ ε, αυξάνεται συνεχώ με υφέρποντα τρόπο η ευρωπαϊκή αρμοδιότητα στα πάντα. Τέλος πάντων, ό,τι και αν αποφασίσουμε τώρα δεν θα κρίνει αυτό την ε, συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Σκέλη. Ε, ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περάσαμε 5-6 χρόνια ασχολούμενοι με το θέμα αυτό. πρώτα απ' όλα με διάφορους άλλους συναδέλφους στο παρελθόν. Χαίρομαι που υπερψηφίστηκε αυτό από τους ε, συναδέλφους ε, και έχουμε άρα αρκετές πιθανότητες να προχωρήσει αυτή η πρόταση και να τελειώσει αυτή η αλλαγή των ρολογιών ε, δύο φορές το χρόνο. Το έτος 2021 θα αποτελεί μια ευκαιρία να εξετάσουμε αυτό το θέμα και να δούμε το κάθε κράτος μέλος αν προτιμά να έχει θερινή ή χειμερινή ώρα. Προσωπικά, εντάξει, κάποιοι όπως ο κύριος Χάναν ε, και εγώ ε, είμαστε υπέρ της ώρας. Νομίζω αυτό θα προτιμάει και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία. Τουλάχιστον σε αυτό να παραμείνουμε ενωμένοι. Σας ευχαριστώ, κύριο Σόσνιερ. Επιτέλους, κάτι που μπορώ να υποστηρίξω. Γιατί επιτέλους μπορούμε να συντάξουμε έκθεση που δεν μιλάει για τα δικαιώματα των λάδων, για την ισότητα των γυναικών, για την ε, διαβίβαση χειρών μηνυμάτων προς τον υπόλοιπο κόσμο και ούτω καθεξής. Επιτέλους αποφασίζουμε κάτι πολύ σημαντικό, όπως την κατάργηση της εποχικής αλλαγής της ώρας. Επιτέλους μπορώ να συμφωνήσω με κάτι και να το υποστηρίξω. Με μεγάλη ικανοποίηση λοιπόν υπερψήφισα τη σχετική έκθεση. Θα πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις ε, αλλαγές εποχικές. Ένα, ε, μην χρειάζεται να αλλάζουμε κάθε τρει και λίγο τα ρολόγια. Δεν χρειαζόμαστε καν ρολόγια. Νομίζω ότι αυτό είναι μία από τις ελάχιστες καλές αλλαγές που πρότεινε το Κοινοβούλιο στην τρέχουσα θητεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σπόλτσακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση για την κατάργηση των εποχικών αλλαγών ώρας και ομολογώ ότι χαίρομαι ιδιαίτερος για την υποστήριξη που επιφύλαξαν στην πρόταση οι Ευρωπαίοι πολίτες και μάλιστα ήταν ε, μία από τις πρωτοβουλίες των πολιτών που προκάλεσαν την άμεση σχεδόν αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χαίρομαι που επιλήθηκε τόσο γρήγορα. Αλλά ο χρονικός ορίζοντας το 2021 νομίζω παρά είναι μακρινός, απόμακρος για πολλούς πολίτες, Ευρωπαίους πολίτες. Ε, Άλλε ήταν οι προσδοκίες των πολιτών να έχουμε πιο άμεση εφαρμογή, πολύ νωρίτερα από τους 18 μήνες. Πάντω είμαι αρκετά ευέλικτο και ελαστικό σε αυτό το θέμα. Μπορώ να δεχτώ τις ε, προτάσεις των εθνικών αρχών ή τη Ευρωπαϊκή Αρχής. Δεν έχω πρόβλημα ούτε με τη χειμερινή ούτε με τη θερινή ώρα. Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτείνεται από την Πορτογαλία προς ε, τις ανατολικές χώρες ή από το Βόρειο Πόλο προ τι νότιε χώρε. Οπότε όντω υπάρχουν διαφορέ. αλλά μπορώ να δεχτώ οτιδήποτε λύση. Ευχαριστώ. Περνάμε στην επόμενη έκθεση, την έκθεση του κυρίου Μπούζεκ για του κοινού κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού. Το λόγο του κύριου Μπενίτο Θιλουάγα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα ψηφίσαμε τη μετερρύθμιση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και επιτέλους αναγνωρίζουμε ε, τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς και τις ε, ενεργειακές κοινότητες ως βασικούς παράγοντες για την ε, μετάβαση την ενεργειακή που δεν θα υλοποιηθεί χωρίς την ανάμειξη των Ευρωπαίων πολιτών και σε έναν εκδημοκρατισμό και μια αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος. Δεν θα πρέπει η ενεργειακή μετάβαση να παραμείνει στα χέρια μόνο των μεγάλων επιχειρήσεων. Θα πρέπει να φέρουμε στο επίκεντρο τον πολίτη, ακόμη και τη ενεργειακή μετάβαση. Θέτουμε όρια στου μηχανισμού ικανότητα και το 2025 έχουμε ε, ανώτατη προθεσμία για, τις, ε, για τα θερμοελεκτρικά εργοστάσια που ρηπαίνουν ιδιαίτερω. Επίσης, θα πρέπει να αποφύγουμε τις ε, και ε, επιδοτήσεις προς ε, ορυκτά καύσιμα ή προς την πυρηνική ενέργεια. Και θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη την κοινωνική επιτακτική ανάγκη να μην αφήσουμε κανένα πολίτη πίσω, να μην περιθωρήσουμε κανέναν και να δώσουμε εναλλακτικέ λύσεις στους εργαζομένους που θα επηρεαστούν από την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Στρογεύσκη. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι πολέμιος α, της υπερβολικής παρέμβασης και της υπερβολικής κανονιστικής ρύθμισης. ε, γιατί μερικές φορές τέτοια υπερβολική ρυθμιστική παρέμβαση δημιουργεί τεράστιο κόστος. Εδώ όμως έχουμε τέσσερις προτάσεις που συμβάλλουν σε κάποιους ελάχιστους κανόνες και προδιαγραφές. Ενισχύουμε τους ε, αποδέκτες, ε, τους καταναλωτές. Δείχνουμε την πρόθεση να ενισχύσουμε την ε, προστασία του περιβάλλοντος, να μειώσουμε τις εκπομπές, αλλά έχουμε μερικές διατάξεις που είναι κάπως προβληματικές. Θα πρέπει επίσης να προβλέψουμε μια επαρκή μεταβατική περίοδο για να μπορέσουν να προσαρμοστούν οι αποδέκτες αυτού του, του κανονιστικού πλαισίου ε, την, για να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες. Η κυρία Κούμπουλα Νάτρη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σημαντική μεταρρύθμιση που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά του κανόνε για την εσωτερική αγορά ηλεκτρική ενέργεια. Μεγάλη ήταν η πλειοψηφία των ε, βουλευτών που υπερψήφισαν την έκθεση αυτή και αποτελεί τελευταία πτυχή τη δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια. Έχουμε λάβει πλέον σημαντικά μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να δημιουργήσουμε μια πραγματική ένωση ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να συμβάλλουμε κατά αυτόν τον τρόπο για την καλύτερη λειτουργία τη αγορά και να έχουμε κατά αυτόν τον τρόπο μια καλύτερη ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και να καταφέρουμε επίση να χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια στο ενεργειακό μείγμα το οποίο προωθούμε. Το μοντέλο λοιπόν αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω της έγκρισης πρότασης αυτής έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Θα μπορούμε πλέον να συνεργαζόμαστε καλύτερα και βέβαια πρέπει να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες στον τομέα αυτό και να είμαστε ακόμα πιο φιλόδοξοι στο μέλλον. Νομίζω θα πρέπει να έχουμε και πιο αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τις εκπομπές. Ευχαριστώ κύριο Σκέλη. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση για τους κοινούς κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως τη σταδιακή κατάργηση των επενδύσεων ε, για, τους, ε, για τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με βάση τον άνθρακα. Θα πρέπει όμως χώρες όπως η Ιρλανδία να έχουν μεταβατική περίοδο για να μπορέσουν να κάνουν την ενεργειακή μετάβαση και περιορισμένες κρατικές ενισχύσεις σε τέτοια, υδροελεκτρικά, ε, σε τέτοια εργοστάσια παραγωγής άνθρακα θα επιτρέψουν την καλύτερη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, μάλιστα το Δεκέμβριο του 2018 είχαμε σχετική νομοθεσία στην Ιρλανδία και παρόμοια πρόταση έχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ορυκτά καύσιμα, κάτι που είναι πολύ ενθαρρυντικό. Βέβαια, ε, εγώ ήμουν ε, εισηγητής για τις ΑΠΕ και θεωρώ ότι οι επενδύσεις της ΑΠΕ είναι επενδύσεις προς ένα πιο καθαρό μέλλον και, μέλλον και ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και χαιρετίζω αυτή την έκθεση γιατί πιστεύω ότι θα διευρύνει την αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προκειμένου να υλοποιήσουμε τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς μας στόχους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Πόλτσακ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η ηλεκτρική ενέργεια και το εμπόριο στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να έχουμε ένα εμπόριο χωρίς φραγμούς, χωρίς εμπόδια, έτσι ώστε ελεύθερα τα κράτη-μέλη να μπορούν μεταξύ τους να εμπλέκονται σε αυτό το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας. Η υπερβολική ρύθμιση θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο, αλλά δεν συμβαίνει ευτυχώς κάτι τέτοιο με την έκθεση αυτή, η οποία νομίζω ότι έρχεται πραγματικά να συμπληρώσει το γενικότερο πλαίσιο, το ενεργειακό, το οποίο προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς υπερψήφισα την έκθεση αυτή, είμαι σαφώ υπέρ της προτινόμενης νομοθεσίας και μην ξεχνάμε ότι αυτό άλλωστε επιδιώκουν και οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ακριβώς την κλιματική αλλαγή θέλουν να αντιμετωπίσουμε, θέλουν να βελτιώσουμε τη θέση των καταναλωτών στα πλαίσια της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και επιθυμούν επίσης οι Ευρωπαίοι πολίτες να υπάρχει ένας ισότιμος ανταγωνισμός ανάμεσα στις διαφορετικές πηγές ενέργειας. Επομένως, χαίρομαι πάρα πολύ για το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα το οποίο εγκρίναμε. Η κυρία Γιαζοβιέτσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν μακροχρόνιες ε, οι συζητήσει για την οδηγία αυτή και ευτυχώ καταλήξαμε σε συμφωνία. Χαίρομαι γι' αυτό. Μεγαλύτερο επίτευγμα της νέας οδηγίας είναι η υιοθέτηση του τρίτου ενεργειακού πακέτου σε όλου τους αγωγού αερίου που, που μεταφέρουν ε, αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης έχουμε υποδομές για την εισαγωγή αερίου από τρίτε χώρε, οπότε νέες, ε, νέ, νέοι αγωγοί θα υιοθετηθούν όπως το Nord Stream 1. Χρειαζόμαστε ε, κοινή πολιτική για την ενεργειακή μας ασφάλεια. Ελπίζω ότι οι νέες διατάξεις θα εφαρμοστούν και στο Nord Stream 2 αγωγό φυσικού αέριου. Ευχαριστώ τον κύριο Μπούζεκ για την θετική του στάση της διαπραγματεύσεις και την ε, μεγάλη του δέσμευση υπέρ του θέματος αυτού και με πολύ ε, χαρά και ακράδαντη υπεποίθηση υπερψήφισα τη σχετική οδηγία. Ευχαριστώ. Περνάμε την επόμενη έκθεση που είναι του κ. Μπούζα και πάλι για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το λόγο κύριο Σέινφελτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι αναφυσβήτητο ότι η εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να αλλάξει θα πρέπει να ενισχυθεί η θέση των παραγωγών ενέργειας στα πλαίσια αυτού του σχεδίου, να επιτρέψουμε διασυνοριακό εμπόριο, να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, να έχουμε φιλοπεριβαλλοντικά μέσα παραγωγής ενέργειας και ε, με καλύτερο περιβάλλον να ε, καταπολεμήσουμε και τις κλιματικές αλλαγές. Για να τα καταφέρουμε όλα αυτά όμως θα πρέπει το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να έχει χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Θα πρέπει ταυτόχρονα να ε, επιταχύνουμε την εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να δώσουμε έμφαση στην αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και ίσως αναμειγνύοντας και τους αποδέκτες ηλεκτρικής ενέργειας, τους καταναλωτές που μπορούν να είναι και παραγωγή ταυτόχρονα. Και φυσικά χρειάζεται κρατική υποστήριξη, δημόσια κονδύλια για το θέμα αυτό. λοιπόν δεν πρόκειται να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Ακριβώς επειδή η έκθεση προσπαθεί να ε, υλοποιήσει όλου αυτού του στόχου, την υπερψήφισε. Ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στην επόμενη έκθεση, πνευματικά δικαιώματα στην ε, ενιαία ψηφιακή αγορά, έκθεση ΒΟΣ. Το λόγο ο κύριος Μαόλου Στέφανο, που φαίνεται όμως ότι απουσιάζει, οπότε περνάμε στην κυρία Μαρίζα Ματίας. Επίσης απουσιάζει, κυρία Γουίντερ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, στην τελική ψηφοφορία πήχα γιατί το αίτημά μου για χωριστή ψηφοφορία απορρίφθηκε για το άρθρο 13. Το δικαίωμα πνευματική ιδιοξίας πρέπει να επιβάλλεται και στον σφιακό κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς αυτό το οποίο τώρα εγκρίναμε ε, μιλάμε για μια αδειοδότηση στο κείμενο αυτό, αλλά εγώ θα προτιμούσα μια καταποκοπή ε, αποζημίωση. Γι' αυτό κατέβηκε τόσο κόσμο στου δρόμου να διαδηλώσει. Γι' αυτό δεν μπόρεσα να συμφωνήσω. Αλλά θεωρώ σωστό ότι θα πρέπει να υποχρεωθούν να πληρώσουν οι πλατφόρμες εκείνες οι οποίες σκοπεύουν να βγάλουν κέρδη με τα όσα ανεβάζονται σε αυτές και βεβαίως να υπάρχει η σωστή διανομή των κερδών. Γι' αυτό δεν μπόρεσα να απορρίψω στο σύνολό τη την οδηγία. Ελπίζω τώρα στην εφαρμογή αυτή τη οδηγία στο εθνικό δίκαιο να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ τη ποικιλομορφία στο διαδίκτυο και προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Σπυράκη, το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα. Ένα βήμα για να δώσουμε την απάντηση ότι η ελευθερία σταματά εκεί που αρχίζει η προσβολή των δικαιωμάτων του άλλου. οι δημιουργοί της ευρώπης οι συγγραφείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να αποζημιώνονται όταν η δουλειά τους χρησιμοποιείται από τις μεγάλες πλατφόρμες. τα πνευματικά δικαιώματα μπορούν να λειτουργήσουν και στην ενιαία ψηφιακή αγορά. οι start up οι πλατφόρμες που τώρα ξεκίνησαν που δεν έχουν χρόνο ζωής περισσότερο από τρία χρόνια που έχουν τζίρο λιγότερο από δέκα εκατομμύρια που έχουν λιγότερους από πέντε εκατομμύρια μηνιαίους επισκέπτες δεν πρέπει να υφίστανται ελέγχους και προδιαγραφές που υφίστανται οι μεγάλες πλατφόρμες. ωστόσο θα πρέπει όλοι να καταβάλουν αποζημιώσεις στους δημιουργούς. οι δημιουργοί είναι εκείνοι που δίνουν νόημα σε όλη αυτή την προσπάθεια. ο ψηφιακό κόσμος οφείλει να διέπεται από κανόνε ακόμη και όταν η ψηφιακή ζωή εξελίσσεται με μεγαλύτερη ταχύτητα από την νομοθεσία εμείς είμαστε εδώ ως νομοθέτες και οφείλουμε να δώσουμε στους πολίτες τα εργαλεία που τους επιτρέπει να προστατεύσουν τη δουλειά τους. σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα καταψήφισα αυτήν την οδηγία. Φοβούμαι ότι το Κοινοβούλιο εδώ πέρα άνοιξε τον δρόμο για μια αντιδημοκρατική μηχανή λογοκρισίας η οποία θα λειτουργεί μόνο με βάση τα οικονομικά ιδιωτικά συμφέροντα χωρίς ε, κανέναν ε, δημοκρατικό έλεγχο. Έτσι δώσαμε στις εταιρείε ΓΚΑΦΑ τη δυνατότητα να λογοκρίνει το διαδίκτυο. Εδώ πέρα καταργείται η ελευθερία γνώμης και βεβαίως η ιδιωτική λογοκρισία θα είναι πολύ ισχυρότερη από όσο ήταν ποτέ η κρατική λογοκρισία δεν ήταν καλή ημέρα σήμερα για τους ε, δημιουργούς ε, είτε στον τομέα της ε, πληροφορικής είτε στον τομέα του περιεχομένου. Μια μαύρη μέρα για το διαδίκτυο. Σας ευχαριστώ κύριε Σόλτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η οδηγία αυτή είναι απαραίτητη. Τη χρειαζόμαστε όλοι, ιδίως οι δημιουργοί, οι συγγραφείς, καλλιτέχνες, εκτελεστές. Σαφώ όμω ε, δεν συνιστά νίκη για κανέναν αυτή η πρόταση οδηγία. και αυτή τη στιγμή από ό,τι φαίνεται τροποποιούμε εντελώ το διαδίκτυο. Γίνεται ουσιαστικά ένα ρομποτικοποιημένο περιβάλλον, αυτοματοποιημένο, όπου τελικό λόγο θα έχουν πάντα οι ε, μεγάλες επιχειρήσει στον τομέα του διαδικτύου μία εβδομάδα ή λίγες μέρες τουλάχιστον μετά την, το πολύ σημαντικό αυτό πρόστιμο το οποίο επιβλήθη στην Google, Εμεί μέσω τη πρόταση αυτή δημιουργούμε περισσότερε ανισορροπίε στην ιστορική αγορά. Το πρόβλημα είναι ο ρόλος που θα έχουν αυτά τα αυτοματοποιημένα φίλτρα, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τελικά πάρα πολύ τα δικαιώματα των χρηστών του διαδικτύου. Και πολύ φοβάμαι ότι η οδηγία αυτή όταν θα αρχίσει να εφαρμόζεται τελικά θα οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα και όχι σε αυτό το οποίο επιθυμούμε. Τελικά θα περιορίσει τη χρήση του διαδικτύου και θα περιορίσει τελικά τη δημιουργικότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριο κύριος έχει το λόγο. Είμαι κατά του συμβιβασμού της οδηγίας ε, copyright λόγω του άρθρου 13 ε, έως 17. Ε, Χαιρετίζω το ότι υπάρχει μια προστασία η οποία προβλέπει αμοιβή για καλλιτέχνε, δημοσιογράφου κτλ. Δεν είναι δυνατόν να παρέχεται δωρεάν η πνευματική ιδιοκτησία. Όποιο το χρησιμοποιεί πρέπει να πληρώνει, αλλά ο έλεγχο μέσω φίλτρων upload είναι κάτι το οποίο μοιραία θα οδηγήσει σε λάθη. Οι αλγόριθμοι διακρίνουν ε, με ανεπαρκή τρόπο το προστατευμένο περιεχόμενο. Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ παλαιού και νέου περιεχομένου, αναλογικού και ψηφιακού. Ελπίζω στην εφαρμογή λοιπόν στα κράτη-μέλη να ληφθούν όλα αυτά υπόψη. Αλλιώς θα περάσουμε σε περιορισμό της ελευθερίας ε, γνώμης. Και θα πρέπει βεβαίως να υπάρχει η πρόσβαση όπως και πριν για όλους. Σας ευχαριστώ κύριε Νέκοφ. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ καταψήφισα τη συμφωνία που προήλθε από τον τριμέρη διάλογο. Δεν θεωρώ ότι η συμφωνία αυτή κάνει σωστή εξισορρόπηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών με τα δικαιώματα των δημιουργών, των δικαιούχων της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χρειάζεται μια μεταρρύθμιση, αλλά όχι ως αυτός σκοπός. Σίγουρα το ευρύ κοινό ε, έχει ήδη ε, αντιδράσει λέγοντας ότι έχουν ε, ξεπεραστεί οι κόκκινες γραμμές και το άρθρο 13 κατά τη γνώμη μου είναι κόκκινη γραμμή. Φυσικά θα πρέπει να βοηθήσουμε τους δημιουργούς και να τους αμείβουμε ανάλογα με, την, με το έργο τους. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να εγγυηθούμε και την ελευθερία. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να υποστηρίξω μια μεταρρύθμιση όπου υπερτερούν τα δικαιώματα του δημιουργού σε σχέση με τα δικαιώματα του καταναλώτη. Ευχαριστώ. Η κυρία Δινόλφη, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξεκινήσαμε με ένα σωστό στόχο, να μεταρρύθμισουμε την οδηγία για τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία, να επικαιροποιήσουμε την οδηγία αυτή μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Και πού καταλήξαμε, εγκρίναμε τελικά ένα κείμενο το οποίο θέτει ένα αμφιβόλο την ελευθερία του διαδικτύου και τα ίδια τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν είναι λοιπόν θετικό το αποτέλεσμα, ιδίω για ανθρώπου σαν και εμένα που είμαι υπέρ τη ελευθερία του διαδικτύου και τη ελευθερία τη έκφραση του διαδικτύου. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε οποιοδήποτε σύστημα το οποίο θα στρέφεται καρτά το δημοκρατικό καθεστώτον. Δεν είναι επιθυμητό λοιπόν το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα άρθρα τα οποία προβλέπουν συγκεκριμένε τροποποιήσει όσον αφορά τις τεχνολογικέ εξελίξει. Αυτά είναι θετικά άρθρα, αλλά από την άλλη έχουμε δύο άρθρα το 11, το 13 και το 10 που στρέφονται κατά των βασικών μα στόχων. Πολύ φοβάμαι ότι τα άθρα αυτά θα θέσουν εν κινδύνο την ελευθερία του διαδικτύου και ιδίω την ελευθερία έκφραση του διαδικτύου. Αυτό είναι απαράδεκτο, κύριε Πρόεδρε. Επομένω, γι' αυτό ακριβώ το λόγο καταψηφίσαμε. Το διαδίκτυο θα πρέπει να παραμείνει ελεύθερο και το κίνημα των πέντε αστέρων θα τάσσεται πάντα υπέρ τη ελευθερία του διαδικτύου. Σα ευχαριστώ, κύριο Μπιουτικόφερ.